Please take Συνεχίζουμε την Ολομέλεια. Αισθάνομαι μια τεράστια χαρά και ευτυχία που βρίσκομαι στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αποκινούμε τις ε, κυρίες συναδέλφους Έξι από αυτές είναι αντιπρόεδροι στο, στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο είναι κοσμήτορες και έχω δίπλα μου και την πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και θα ήθελα συνεχίζοντας τη Σύνοδο της Ολομέλειας να πω ότι εορτάζουμε την εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Θα ξεκινήσουμε με ένα με μια σύντομη ταινία που συνοψίζει την ιστορία αυτής της εξαιρετικά σημαντικής ημέρας. Ας αρχίσει η προβολή παρακαλώ.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 Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, δύο λεπτά ταινίες φυσικά δεν μπορούν να δείξουν όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 100 χρόνια. Πάρα πολλά, χρόνια, πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και αλλού. Πάντω, σε σχέση με άλλε χώρε του κόσμου, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε όμω ότι δεν φτάσαμε στο τέλο τη πορεία μα. Όλο, δυστυχώς έχουμε ακόμη πολύ λίγες γυναίκες στην πολιτική. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μόνο 35% των γυναικών. Βέβαια, το ποσοστό αυτό είναι λίγο υψηλότερο από ότι στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά δεν έρχεται αυτό το 35% της συμμετοχής των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευτυχώς, ε, στις ε, ηγετικές θέσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε άνω το 40% γυναίκες. Και μάλιστα έχουμε και προέδρους επιτροπών. Και έχουμε αρκετές γυναίκες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα γίνει όμως την επόμενη τριετία, μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογέ. Πολλά πράγματα εξαρτώνται και από τα εθνικά κοινοβούλια και από το πώς θα αναδειχθούν ε, οι εκπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να φροντίσουν και να μεριμνήσουν για να αυξηθεί ο αριθμός των ε, γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και απευθύνουμε έκκληση σήμερα, απευθύνουμε έκκληση προς τους συναδέλφους μας από τα εθνικά κοινοβούλια να θεσπίσουν ε, τις απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις και να λάβουν τις αποφάσεις ώστε να αυξηθεί ε, η συμμετοχή των γυναικών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να είμαστε και υπόδειγμα σε ό,τι αφορά την πρόσληψη των γυναικών. 59% των γυναικών, 59% των ε, υπαλλήλων είναι γυναίκες και άνω του 50% είναι επίσης γυναίκες που ασχολούνται με πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Έχω και ίδια εμπειρία από το θέμα αυτό και μάλιστα όταν ήμουν πρωθυπουργός στη χώρα μου είχαμε περίπου 50% των γυναικών στις πιο σημαντικές υπουργικές θέσεις και στις ηγετικές θέσεις σημαντικών κρατικών οργάνων. Και αυτό είναι ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί έκτοτε. Επίσης, ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέφθηνα έκκληση για να αυξηθεί ο αριθμός ε, της συμμετοχής των γυναικών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στις ηθήνουσες και ηγετικές θέσεις της Ένωσης. Και μπορούμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή μας, γιατί είπατε εκπρόσωπος ε, εξωτερικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γυναίκα. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τι ηγετικέ θέσει. Και αυτό θα ευνοήσει όχι μόνο τι γυναίκε, αλλά θα είναι προνόμιο και θα ωφελήσει τι ίδιε επιχειρήσει. Και θα πρέπει να φροντίσουμε, ότι να, θα φροντίσουμε να εξασφαλιστεί η ισότητα των μισθών για τι ίδιε εργασίε. Εφόσον άνδρες και γυναίκε έχουν τα ίδια προσόντα και επιτελούν την ίδια εργασία, θα πρέπει να απολαμβάνουν και τον ίδιο μισθό. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε ακόμη κάποια πρόοδο. Επίσης, πρέπει να δώσουμε μάχη για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα εδώ να αποτίσω φόρο τιμής σε όλες σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Και αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια σκέψη για τις γυναίκες που στην Αγγλική Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική δίνουν τη μάχη τους υπέρ της δημοκρατίας. Α μην ξεχάσουμε και όσους ε, βραβεύθηκαν με το βραβείο Ζαχάροφ, ιδιαίτερα τις γυναίκες, την κυρία Ονσανσουκή, τη Λέιλα Λαζάνα και την Τένα Σελμπλάνκο που βραβεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε καμία περίπτωση και στο όνομα κανένα πολιτικού συστήματο οι θρησκείε δεν θα πρέπει να θυσιάζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν θα πρέπει που δεν είναι και για κανένα λόγο οι γυναίκε στον κόσμο να έχουν λιγότερα δικαιώματα από του άντρε. Θα πρέπει να εκφράσουμε μια φωνή διαμαρτυρία όπου διαπιστώνουμε τέτοιε καταστάσει. Στι 3 Νοεμβρίου, ε, πριν από 200 χρόνια, στην Ευρώπη, Ε, είχαμε την ε, κατάρτιση της διακήρυξης ε, των, γυναικών και των, των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συντάκτρια δολοφονήθηκε. Χρειάστηκαν να περάσουν χρόνια για να αναγνωριστεί το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Και μάλιστα η πρώτη χώρα που κατοχύρισε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες ήταν η Φιλανδία. Μέσα σε 100 χρόνια σημειώσαμε σημαντική πρόοδο ό,τι αφορά την ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά. Η 8η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Αλλά αυτή ε, η γιορτή θα πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι και τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου να μην ξεχνούμε, να θυμόμαστε συνέχεια ότι το πιο σημαντικό σήμερα ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ισότητα ανδρών και γυναικών. Και καθ' όλη τη διάρκεια του έτου, ε, σε όλε αυτέ τι 365 μέρε θα πρέπει να ισχύουν οι αρχέ που τιμούμε την 8η Μαρτίου. Δεν αρκεί να έχουμε μία μόνο μέρα, δεν αρκεί η 8η Μαρτίου. Θα πρέπει και τι υπόλοιπε μέρε του χρόνου να έχουμε κατά νου το ίδιο θέμα, το θέμα τη ισότητας ανδρών και γυναικών. Σα ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στις συναδέλφου. εκ μέρου Συμβουλίου στην κυρία Νίκο Γκιόρη την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο, κυρία Γκιόρη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Επιτρέψτε μου να σας απευθύνω το λόγο στη μητρική μου γλώσσα σε αυτή την επαιτειακή συνεδρίαση. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ε, την πρώτη φορά που ε, ακούστηκε αυτή η ιδέα ήταν επαναστατική ότι οι άνδρες είναι ε, ίση με τις γυναίκες και έχουν οι γυναίκες τα ίδια δικαιώματα. Ε, είναι θέμα αξιοπρέπειας, ίσης αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, δεν αρκεί η απλή έκδοση διακηρύξεων. Καμιά φορά διαφέρουν οι καταστάσεις και ως προς τη γυναική αξιοπρέπεια από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αυτές οι ε, πετειακές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα ε, αμέσως μετά τη συζήτηση που είχαμε για τη γυναική αυτόχεια. Η οικονομική κρίση πλήττει ε, περισσότερο τις πιο ευάλωτες ομάδες και μεταξύ αυτών είναι και οι γυναίκες και πραγματικά αυτό μας αναγκάζει να αντιδράσουμε. Ναι, επιπλέον, ε, τα προβλήματα αυτά είναι κάτι που αφορούν ε, τον κόσμο ολόκληρο, όχι μόνο ε, την Ευρώπη. Ακούμε συχνά ότι η φτώχεια έχει γυναικείο πρόσωπο οι γυναίκες ε, πολλές φορές χρειάζεται να ε, ξεφεύγουν από ε, πολέμους σε συνθήκες φτώχειας, με παιδιά, χωρίς άνδρες και μεταξύ της των προτεραιοτήτων συγγνώμη, της Ουγγρικής Προεδρίας είναι πολλά θέματα που αφορούν την πρόθεση της εργασίας των γυναικών. Στη στρατηγική ε, Ευρώπη 2020 έχουμε στόχους και για την απασχόληση που θα συνεισφέρουν ε, στη μείωση της φτώχειας. Η απασχόληση των γυναικών αναφτερώνει την αξιοπρέπεια των γυναικών, τους επιτρέπει ε, να αποφασίζουν και να ζουν ελεύθερα. Η εμβληματική πρωτοβουλία, η πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας, επίσης ε, τονίζει και αναδεικνύει τη σημασία των διαφορών ε, ε, μεταξύ των συνθήκων απασχόληση ανδρών και γυναικών. Είναι σημαντικό επίτευγμα η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ισότητας των Φύλων δεν θα πρέπει να λησμονούμε τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες οι οποίες καλούνται να συγκεράσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό τους βίο και ε, θα πρέπει να μπορούν να το πράττουν με ελευθερία επιλογής. Επίσης προβλέπουμε μια οδηγία για τη βελτίωση ε, των συνθηκών εργασίας ε, των εγγύων γυναικών ή των μητέρων σε περίοδους λοχίας και θυελασμού. Επίσης διοργανώνουμε ε, τη Εβδομάδα Δημογραφίας με ε, συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς επίσης και Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων με στόχο να συζητήσουμε μέσα και τρόπους αύξησης των γεννήσεων στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες ε, μειονεκτούσες περιμένουμε από το Συμβούλιο να εγκρίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στρατηγική υπέρ το Ρωμά τον Ιούνιο. Η κυρία Γιάροκα και άλλοι βουλευτές εδώ συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή και θα ήθελα να τονίσω και το ρόλο των γυναικών στις κοινότητες των Ρωμά ε, ε, πώς εξασφαλίζουν την οικογενειακή συνοχή. Είναι σημαντικός ο ρόλος τους και ένα τελευταίο. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι χωρίς ενεργή κοινωνική συμμετοχή των γυναικών δεν νοείται ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Εσείς ο ίδιος πρόεδρε αναφερθήκατε σε γυναίκες που απαιτούν ε, την ελευθερία του στην πλατεία Ταχρήρ του Καΐρου. Και αυτές οι γυναίκες θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το μέλλον τους οι προσπάθειές τους και αγώνες τους θα πρέπει να υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με γενοδορία, ανοιχτά και ειλικρινά, χωρίς ιδεολογικά στερεότυπα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Προεδρεύουσα. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον κύριο Μπαρόσο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να πει και εκείνος δύο λόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σήμερα θυμόμαστε τις φωνές εκείνων των γυναικών που στις 19 Μαρτίου του 1911 ξεκίνησαν από τη Γερμανία, τη Δανία, ε, την Ελβετία και την Αυστρία και ένωσαν τις φωνές τους ε, για να υπερασπιστούν τις γυναίκες και τις ε, συνθήκες εργασίας. Ο πρόεδρος διακόπτη τον κύριο Μπαρόσο. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε ησύχως και χωρίς συζητήσεις στο ημικύκλιο. Είμαστε σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση. Παρακαλώ συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Μπορείτε να αρχίσετε ξανά. Αν Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, λέει ο κ. Σήμερα τιμούμε ένα αιώνα αγώνων και επιτυχών αγώνων από τους οποίους έχουμε υποφεληθεί όλοι. Τι θα ήταν άραγε οι δημοκρατίες μας και ιδιαίτερα η δημοκρατία στην Ευρώπη που εδώ στο Κοινοβούλιο εκπροσωπείται χωρίς την πλήρη και ε, ε, αμέριστη συμμετοχή των γυναικών ποια θα ήταν η ποικιλομορφία μας, η διαφορετικότητα, ποια θα ήταν η κοινωνία μας και η οικονομία μας χωρίς το ταλέντο των γυναικών. Πολλές φορές οι ε, Ευρωπαίες γυναίκες είναι πρότυπα για τον υπόλοιπο κόσμο από πολλές πλευρές. Η θέση που καταλαμβάνουν οι γυναίκες στην κοινωνία μας είναι πηγή έμπνευσης για γυναίκες απανταχού της γης. Θα ήθελα υπό την έννοια αυτή εδώ να αναφερθώ στο θαραλέο αγώνα των γυναικών της Βορείου Αφρικής που στο πλευρό των ανδρών κάνουν τώρα ό,τι μπορούν για να αντισταθούν στις δικτατορίες και να εγκαθιδρύσουν δημοκρατίες. La Η ενεργή θέση που ε, καταλαμβάνουν σήμερα οι γυναίκες στην οικονομική και πολιτική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα της ε, ε, στεναρής τους δέσμευσης και στράτευσης και χαιρετίζουμε ε, ε, μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ισότητα ε, ανδρών και γυναικών και κατοχυρώνεται πλήρως στη συνθήκη της Λισαβόνας. Κατά τη διάρκεια των ετών, μια σημαντική νομοθεσία για την ισότητα των αμοιβών και την ένταξη του φύλου στις ευρωπαϊκές πολιτικές επέτρεψε να προχωρήσουμε προς μια κοινωνία με μια αγορά εργασίας πιο ίση. Θα πρέπει όμως να αγανακτούμε ακόμα και σήμερα για αυτά που παραμένουν ε, απογοητευτικά και απαράδεκτα. 62,5% ε, είναι ο μέσος όρος εργασίας των γυναικών, ενώ στους άνδρες είναι 80%. Όλο και μεγαλύτερη επιτυχία στην εκπαίδευση των γυναικών έρχεται όμως σε σύγκρουση με τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Αυτό παραμένει απογοητευτικό και θα πρέπει να αλλάξει οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε ε, χαμηλόμιστες και επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και υποαπασχολούνται σε θέσεις ευθύνης. Διαφορά επίσης αμοιβή ανδρών και γυναικών της τάξης του 18% παραμένει και μεταφράζεται ε, σε κίνδυνο για 22% των γυναικών ηλικίας άνω των 65 ετών να πέσουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας γιατί δεν έχουν αρκετή σύνταξη και αυτό είναι επίσης απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 με 25% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστεί ε, σωματική βία τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Και αυτό επίσης είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει. Σήμερα θα πρέπει να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού έτσι ώστε η ισότητα ανδρών και γυναικών να γίνει πλήρης πραγματικότητα. Έχουμε να κερδίσουμε όλοι από αυτό. Είτε πρόκειται για κοινωνική και οικονομική συνοχή, η φόρο ανάπτυξη, είτε ανταγωνιστικότητα. Το Σεπτέμβριο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική με πέντε τομείς δράσης προτεραιότητας για την περίοδο 2010-2015. Ισότητα στην αγορά εργασίας και οικονομική ανεξαρτησία εξίσου για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ισότητα μισθών. Ισότητα στις θέσεις ευθύνης προώθηση της ισότητας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πάντα στο πλευρό των γυναικών που ε, ανά τον κόσμο αγωνίζονται καθημερινά για να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην εργασία, για γυναίκες που αγωνίζονται για τον εκδημοκρατισμό και την άσκηση των ελευθεριών και των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι ε, περνάει από το χέρι για να ε, συνεισφέρει στην εκπλήρωση αυτών των στόχων. Αλλά ας μην λησμονούμε ότι οποιαδήποτε νομοθεσία όσο καλά και αν εφαρμόζεται δεν πρόκειται να λύσει τα πάντα. Τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις που θα πρέπει επίσης να αλλάξουν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα εορτάζουμε τον αγώνα των γυναικών για την ισότητα. Σήμερα μπορούμε να πούμε στην Ευρώπη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν αδύνατη χωρίς τις Ευρωπαίες, όλες τις Ευρωπαίες. Είναι ουσιαστικότατη η συμμετοχή τους ε, στο κοινό μας εγχείρημα που βασίζεται στις αξίες μας και συμμελαμβάνει μεταξύ αυτών και την ισότητα ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ. Η κυρία Εύα Μπρίτς Βένσον, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Διοφύλων και Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Yeah. Okay. Man eh, föds inte till kvinna, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η γυναίκα δεν γεννιέται κανείς, αλλά γίνεται αυτή η σημαντική ρίση αποδεικνύει ε, ποιες είναι οι απόψεις ε, των ε, ανδρών και ποιες είναι οι επιλογές μας. Επιλογές βασίζονται περισσότερο στο φύλλο και όχι στις δεξιότητές μας. Τα στερεότυπα για τα δύο φύλλα υπάρχουν στους άντρες και τις γυναίκες και τα 100 χρόνια αγώνα για την ισότητα δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν αυτά τα στερεότυπα. Αλλά όμως εμείς δεν θα περιμένουμε άλλα 100 χρόνια, ακριβώς διότι υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα για τα δύο φύλλα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το 97% των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων διευθύνονται από άνδρες. Οι γυναίκες ε, καλύπτουν, ε, αν έχουν δουλειά, τις περισσότερο ανασφαλείς θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες είναι εκείνες ε, οι οποίες εργάζονται στο σπίτι χωρίς αμοιβή. Οι γυναίκες είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο φέρουν την ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών. Οι γυναίκες είναι θύματα βίας, είναι εκείνες που είναι πολλές φορές θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων είναι οι γυναίκες που στο εμπόριο γυναικών ε, πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως ε, αντικείμενο, ως αγαθά. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις ε, κοινωνίες μας υπάρχουν ε, διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Σίγουρα ε, έχω υπάρξει πρόοδο τα τελευταία 100 χρόνια γιατί συγκρίνω τις ευκαιρίες που είχα εγώ παραδείγματος χάρη με τις ευκαιρίες που είχε η μητέρα μου και αν θέλετε και η αγιά μου και πράγματι καταλήγω στο ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος. Όμως υπολείπουν ακόμα πάρα πολλά και γι' αυτό ο αγώνας συνεχίζεται κάθε ημέρα του χρόνου και όχι μόνο στις Μαρτίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Λίδια Γιαρόκα. Ευχαριστώ. Εορτάζουμε την εκατοστή υπέτειο της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Μάλιστα το 19ο αιώνα οι γυναίκες εργαζόμενες ζήτησαν ίσο μισθό για ίση εργασία. Αυτό συνέβη το 1957, πριν από 50 χρόνια και. Αλλά εξακολουθεί δυστυχώς να είναι έγκυρος αυτός ο στόχος, ε, γιατί οι γυναίκες ε, κερδίζουν 15% λιγότερο από τους άνδρες για ίση εργασία και στην ε, Ουγγαρία πάνω από 16%. Και παρόλο που η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού είναι γυναίκες, οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 10% του παγκόσμιου πλούτου. Είναι τεράστιο το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, δυστυχώ ακόμη. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τα δικαιώματα των γυναικών. Άλλωστε, οι γυναίκε είναι πιο ευάλωτε ε, απέναντι στη φτώχεια. Το γεγονό ότι κάποια γυναίκα είναι μόνη τη με παιδί θα πρέπει να την φέρνει πιο κοντά στη φτώχεια και να την εκθέτει περισσότερο σε περιθωριοποίηση. Δυστυχώ δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών στην εργασία σε πολλέ ε, περιοχέ ακόμη. Όχι μόνο του κόσμου, αλλά και τη Ευρώπη και γίνονται και θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τα φαινόμενα κακής μεταχείρισης και οικιακή βίας ε, εις βάρος των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, ας μην γίνονται συζητήσεις εντός της Επόμενο Επόμενος ομιλητής εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Μπρίτα Τόμσον. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από 100 χρόνια για πρώτη φορά ε, έλαβε χώρα η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και τι ζητούσαν τότε. Το, ε, εκλογικά δικαιώματα. Για σήμερα είναι τελείω φυσικό και αυτονόητο αυτό. Χρειάζεται όμω να διανύσουμε πολύ δρόμο μέχρι την πλήρη ισότητα. Και θα ήθελα να τονίσω πραγματικά ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι γυναίκε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Και στην πολιτική αλλά και στην οικονομική ζωή. Οι γυναίκε επίση θα πρέπει να είναι παρούσε στι τράπεζε δεν είναι δυνατόν ο μισός πληθυσμός να αποκλείεται από τις σημαντικές οικονομικές ε, ε, θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλο το ταλέντο του πληθυσμού και ε, των γυναικών και αυτό είναι σημαντικό και για την ανταγωνιστικότητά μας. Γι' αυτό και καλωσορίζω την πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ. Είναι πάρα πολύ θετική. Ακριβώς και εν ώψη της υλοποίησης της ισότητας. Χρειαζόμαστε περισσότερα από απλώς μια συμβολική πολιτική και ελπίζω να έχουμε αυτό το θάρρος. Επόμενη ομιλήτρια εξ ονόματος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, η κύρια Αντιπρόεδρος Σιλβάνα Κοχμερίν. Herr Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, στην ε, διακήρυξη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων τα δύο πρώτα άρθρα αναφέρονται στην ισότητα όλων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και γεννιούνται με αξιοπρέπεια έχουν ε, λογική νου και πρέπει να συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλον με αδελφικό πνεύμα. Θαυμάσια αυτή η αναφορά, όμως 100 ε, χρόνια μετά την ε, πρώτη επέτειο περί της ημέρας των γυναικών δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απόλυτη ισότητα. Σίγουρα στην Ευρώπη έχουμε επιτύχει πάρα πολλά και σήμερα αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι κυρίως η νομική ελευθερία της γυναίκας γιατί αυτήν την έχουμε κατοχυρώσει σε μεγάλο βαθμό. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις φεμινίστριες των περασμένων ετών για όλα αυτά που έκαναν για μας. Σήμερα αυτό που ενδιαφέρει είναι η ελευθερία που βιώνουμε. Οι άνδρες πρέπει να δεχτούν τον συμβιβασμό της οικογένειας με τη δουλειά, το πώς μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν, να δεχθούν ότι είναι αυτονόητο οι γυναίκες να είναι πρωθυπουργοί ή υπουργοί. Και είναι θαυμάσιο το να βλέπει κανείς ε, πώς ε, οι γυναίκες ε, στην Αφρική έχουν το βλέμμα στραμμένο σε εμά. Σε εμά γιατί εμείς καλούμεθα να διαδραματίσουμε το ρόλο του σκαπανέα. Δεν πρέπει λοιπόν να χάνουμε το στόχο από τα μάτια μας. Ο στόχος είναι να βιώνουμε την ελευθερία. Γιατί μόνο τότε η ισότητα των δύο φίλων θα είναι κάτι το αυτονόητο και η Διεθνή ημέρα των γυναικών από απλή επέτειο θα είναι μια πραγματική ημέρα ελευθερίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ε, ομιλητρία εκ μέρους των Πρασίνων, αντιπρόεδρος ε, κυρία Κράπη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι τέτοια που δεν καλεί για επαιτειακά πανηγυρικά ε, ε, σχόλια και εορτασμούς. Ακριβώς την εκατοστή επέτειο ως γυναίκες εμείς θα πρέπει να στραφούμε στο παρελθόν και να βγάλουμε έναν απολογισμό. Ο δικός μου απολογισμός είναι ότι η ίση μεταχείριση θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένη και ε, διατρανωμένη σε νομοθεσίες και συντάγματα. Εντάξει, για να γίνει πραγματικότητα όμως θα πρέπει να έχουμε και καθημερινούς νόμους που να εφαρμόζονται. Και εκεί ανήκει για μένα η ποσόστοση. Ας κοιτάξουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη από ό,τι στην κορυφή των ε, οικονομικών επιχειρήσεων. Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις πραγματικά στην κορυφή είναι σπάνιες. Και για να το επιτύχουμε αυτό κυρία Ρέντιν και κύριε κύριε Μπαρόζο, χρειαζόμαστε μια ε, πραγματική σκληρή ρύθμιση ποσοστώσεων και θα χαιρόμουν αν είχατε βγάλει ένα τίμιο, ένα ειλικρινή απολογισμό για τη μη ίση μεταχείριση των γυναικών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γιατί έτσι θα ξέρατε πόσο απαραίτητη είναι αυτή η ποσόστοση. Σήμερα κατά την άποψή μου είναι έσχος, είναι ντροπή το γεγονός ότι οι γυναίκες με πολύ μεγάλα προσόντα και οι δεν έχουν ακόμα χώρο εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσει σε ηγετικό επίπεδο και τίθεται τα θεμέλια της πολιτική. Η ποσόστοση είναι το απαραίτητο όργανο και κυρία ε, Ρέντινγκ αυτή την εκατοστή επέτειο το ζητούμε από εσά. Δεσμευτείτε παρακαλώ ότι θα φέρετε πραγματική ποσόστοση για τι γυναίκε ηγετικέ θέσει, όπω ισχύει άλλωστε στην Νορβηγία και τώρα ήδη και στην Ισπανία και στη Γαλλία να εφαρμοστεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ε, το ανέφερε στην ομιλία του κάνω ο κύριος Μπαρόσο. Ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη εκ μέρου των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Την περασμένη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασιλείο, ο Λόρδο Ντέβι έκανε την ομιλία του προ την κυβέρνηση για την αύξηση τη συμμετοχή των ε, γυναικών και μάλιστα έχει κάποιους ε, προαιρετικού στόχου για τι επιχειρήσει. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες, αλλά δεν ε, χρειαζόμαστε ποσοστό για κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό είναι πατροναριστικό. Το ίδιο με, την, ε, με το τριαντάφυλλο που μας δώσετε μπαίνοντα στην αίθουσα. Προτιμώ να δώσω το δικό μου τριαντάφυλλο σε έναν άνδρα. Εν πάση περιπτώσει και πιο θετικά, νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία μειώνει το χάσμα το μισθολογικό μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχει μειωθεί, ε, κατά 10, έχει μειωθεί στο 10% το χαμηλότερο χάσμα από τότε που διαπιστώθηκε αυτό το φαινόμενο. Επίση, θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στη μητρότητα. Γιατί η πραγματική ισότητα είναι και το δικαίωμα επιλογή και καμία κρίση για την επιλογή. Γιατί όταν, ε, όταν κάποια γυναίκα. Ε, έχει προβλήματα και δεν μπορεί να κάνει την επιλογή της, τότε δεν υπάρχει ελευθερία. σε όποιο στρώμα και είναι και αυτή η γυναίκα, ό,τι δουλειά και αν κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χίλντα Φιγκερέντο, εκ μέρους της Ενωμένης Αριστεράς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε τον αγώνα των γυναικών για την ελευθερία, για την κοινωνική πρόοδο και για την ειρήνη. Μια στιγμή που εορτάζουμε και την εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Ήταν πολλοί αγώνες και πολλές οι κατακτήσεις που επέτυχαν οι γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της εκατοντήρης Αλλά δεν ήταν αρκετές αυτές οι μάχες και οι επιτυχίες για να αρθούν όλες οι ανισότητες και όλες οι ανισορροπίες οι μισθολογικές ανισότητες, οι ανελαστικές μεταρρυθμίσεις, η δυσκολία τους να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία τους και η δυσκολία πρόσβασης σε ε, ηγετικές θέσεις ή σε θέσεις ε, πολιτικής ευθύνης. Και μάλιστα η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται εν μέσω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Και η μητρότητα παρόλο που είναι σημαντική κοινωνική λειτουργία και απαραίτητη για την εξέλιξη της κοινωνίας οι γυναίκε υφίστανται διακριτική μεταχείριση όταν είναι μητέρες και εργαζόμενες ταυτόχρονα. Κάτι που πραγματικά είναι σκανδαλώδες στον 21ο αιώνα. Θα πρέπει να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη τη ομάδα μας προς τον αγώνα των γυναικών και να απαιτήσουμε να τεθεί ένα τέρμα στις ανισότητες και τις διακριτικές μεταρρυθμίσεις και στην γενικευμένη βία εις βάρος των γυναικών. Θα πρέπει να καταργηθούν τα στερεότυπα για τα δύο φύλλα και να περάσουμε από τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ, σε εναλλακτικέ πολιτικέ που θέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ενισότητα των δύο φύλων στο επίκεντρο τη λήψη των αποφάσεων και στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών. Σα ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Μάρα Μπιτσότο, εκ μέρου τη Ευρώπη Ελευθερία και Δημοκρατίας. Πολλοί εξημών, ε, πολλά έχουν επιτευχθεί, ακόμα όμως ε, ε, πρέπει να έπονται πολλές μάχες. Οι γυναίκες βρίσκονται μέσα σε διαμάχες. Είναι δύσκολο λοιπόν να διεκδικήσουμε ελάχιστα μέτρα της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς. Ε, δεν μπορούμε να εορτάσουμε σήμερα την ημέρα της γυναίκας χωρίς να έχουμε στραμμένο το βλέμμα στις μουσουλμάνες γυναίκες ε, στις, στις, ε, στην Αφρική και στις αραβικές χώρες. Είναι δικό τους πρόβλημα, σύντομα όμως θα γίνει και δικό μας. Και δεν μπορούμε να αγνοούμε τους αριθμούς που κάθε χρόνο δίνουν αύξηση. αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που και που έχουν παιδιά που βρίσκονται στα δικά μα τα σχολεία. Οι ίδιε οι μουσουλμάνε γυναίκε αντιμετωπίζουν τη βία στην οικογένειά του. Εγώ εδώ και καιρό ζητάω η Ευρώπη επιτέλου να εφαρμόζει μια στοχευμένη πολιτική για το πώ μπορεί να εξαλειφθεί ο ακραίο φανατισμό στι μουσουλμανικέ χώρε. Να υπάρχει αξιοπρέπεια τη γυναίκα, να μην υπάρχει βία κατοίκον βία. Εμεί οι Ευρωπαίε γυναίκε πρέπει να αγωνιστούμε για εκείνε που ζουν στην Ευρώπη αλλά ε, έχουν, τους έχει αφαιρεθεί η φωνή από τον ε, φανατικό Ισλαμισμό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νικόλ Σενκλέρα, από τους μη γεγραμμένους. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αποτίσω ένα φορό τιμή σε όλες τις γυναίκες, σε όλο τον κόσμο και ε, όχι μόνο τα 100 τελευταία χρόνια αλλά και παραπάνω που έχουν αγωνιστεί για την ισότητα. Βεβαίω το 1893 έδωσε η Νέα Ζηλανδία δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες και επιπλέον το 1970 ε, η Μπάρμπαρα Κάρσο έφερε τον πρώτο νόμο ε, για την ίση αμοιβή. Ε, και επίσης ήμασταν η πρώτη χώρα που είχαμε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό. Πρέπει να το πω και αυτό για τη χώρα μου, στην Ευρώπη. Ωστόσο η Ευρώπη σήμερα έχει χάσει την επαφή της με την πραγματικότητα. Εγώ είμαι κατά των διακρίσεων, πάσης φύσεως, ακόμα και των θετικών γιατί αναπόφευκτα αυτό οδηγεί ε, στην ύπαρξη θυμάτων. Δεν χρειάζεται οι γυναίκες να ε, πατρονάρονται, να χειραγωγούνται ε, από ποσοστώσεις. Τα κράτη-μέλη καλά θα κάνουν να βελτιώσουν τη φροντίδα και τη φύλαξη των παιδιών. Με παρόλη τη θέση της Ευρώπης ε, για τη θετική διάκριση υπέρ των γυναικών δεν συμφωνώ. Χρειάζεται ε, κάτι που να μην κάνει τη ζωή των γυναικών πιο ακριβή και πιο δύσκολη. Ε, Ολοκληρώνουμε την πανηγυρική μας συνεδρίαση και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ.